έχουμε τις παρεμβάσεις διαρκές ενός λεπτού. Πρώτη θα λέει το λόγο η κυρία Κλούνα. Έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω για το θαλάσσιο περιβάλλον και πόσο σημαντικό είναι για τις ε, κοινότητες της ε, υπαίθρου. Όλα αυτά τα οποία είπαμε σήμερα για την Αιλία είναι προ όφελο αυτών των αγροτικών κοινοτήτων. Και πέρυσι, δεν είχαμε πει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Κόρκο που είχε γίνει μια διάσκεψη σε σχέση με την γαλάζια η οικονομία, η ισχυρή ανάπτυξη και όλα αυτά τα βάλουμε υπόψη στην Ιρλανδία και προσπαθούμε αυτά να τα να φυτεύσουμε στην οικονομία σε να την πολλιάσουμε με αυτά και για κάθε 100 ευρώ που παράγονται από την γαλάζια οικονομία τα 75 με 80 πηγαίνουν σε άλλους συναφείς τομείς και μιλάμε ότι αυτό έχει σχέση με την μεταποίηση, την ε, αλία, έρευνα, καινοτομία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Επίτροπος, ξέρω ότι έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν την ε, γαλάζια οικονομία και έτσι να στηρίξουν τις αγροτικές περιοχές και τις αγροτικές κοινότητες. Next one, Mr. Negrescu. επόμενη. Ο κύριος Νεγκρέσκου, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θέλουμε να υπάρχουν κάποιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Να υπάρχει ισότητα. Αυτό το καταφέρει η αγορά. Αυτοί οι οποίοι κρύβουν τα χρήματά τους στους φορολογικούς παραδείσους πρώτα-πρώτα είναι ανήθικοι. Πέραν αυτού όμως. Ο τύπος στην ε, Ρουμανία αναφέρει ότι τα ποσά τα οποία πήγαν στους φορολογικούς παραδείσους αντιστοιχούν στον προπολογισμό της υγείας στην χώρα μας. Θα πρέπει να υπάρξει ελληνικός μηχανισμός, φορολόγηση, να υπάρξουν αυτοί οι μηχανισμοί για να μπορέσουμε να παρέμβουμε. Σας υπενθυμίζω ότι πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες έχουν εγκρίνει τον φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Η κυρία είναι η επόμενη μαγκλήτρια. Ε, το δικαστήριο της ε, Χάγης ε, καταδίκασε τον κύριο Σέτσελη. Δεν καταδίκασε το Σέσελ, ο οποίος ήταν υπεύθυνο για τα σημαντικότερα εγκλήματα του πολέμου. και αυτό αντιβαίνει σε άλλες αποφάσεις του ίδιου δικαστηρίου. Όποιος είναι εξοικειωμένος με την πρόσφατη πολιτική ιστορία και τα συμβάντα τη δεκαετία του 1990 στη Ιουγκοσλαβία γνωρίζει ότι η Κροατία και η Σερβία δεν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με άλλο τρόπο. Άρα λοιπόν η απόφαση αυτή όχι μόνο ε, υπονομεύει τη διαδικασία συμφιλίωσης αλλά και το διεθνές δίκαιο. Μετά από αυτή τη δίκη πολλές ε, χώρες δεν θα θέλουν να συνεργαστούν με τα διεθνή δικαστήρια και αυτό θα έχει ένα αρνητικό αντίκτυπο στην ειρήνη και τη σταθερότητα στον κόσμο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την 30η επέτειο της καταστροφής του πυρηνικού σταθμού της στην Ουκρανία, του Τσερνόμπιλ. Έγιναν σημαντικές προσπάθειες ανάκτησης και βεβαίως έχει μετρηθεί, έχουν μετρηθεί πολύ ψηλότερα ποσοστά καρκίνου ανάμεσα στους εργαζόμενους ο κανονισμός άλλαξε το 2003 που προέβλεπε ε, παροχές και έκτοτε μόνο αν έχει κάποιος αναγνωριστεί ως παθόν έχει δικαίωμα, έχει δικαίωμα σε παροχές. Ο περιορισμός αυτός αφορά ε, συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμών. Αγαπητοί συνάδελφοι, η έμεση διάκριση αυτών που έχουν ε, υποστεί βλάβη από το ε, ατύχημα του Τσερνόμπιλ θα πρέπει να σταματήσει. Σας ευχαριστώ. And now, Mrs. Albiol Guzman. Ευχαριστώ πολύ. Η οικογένεια στην οποία συγκαταλέγεται ο Επίτροπος κ. Κανιέτε έχει λάβει μεγάλα ποσά που αφορούν την ΚΑΠΑ. Αυτό θα ήταν επαρκές, επαρκές λόγο, λόγος να εμφανιστεί ο κύριος Κανιέτε στο Ευρωκοινοβούλιο γιατί ε, και, και εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι η κυρία Μικαέλα Ντομέκ είναι μια από τις ε, ε μία από τις οποίες κατηγορούνται και το όνομα της εμφανίζεται στα, στα κείμενα στα Panama Leaks. Ε, κύριε Κανιέτε, επιτέλους ε, παρετηθείτε. Ευχαριστώ πολύ το Δεκέμβριο ε, ε, του 1991 η μεγαλύτερη πλειοψηφία, του Καραμπάχα ε, ψήφισε για την ανεξαρτησία. Ωστόσο ο πόλεμος με το Αζερβαϊτζάν ε, προκάλεσε πάρα πολλούς ε, θανάτους. Η δημιουργία της ομάδας του Μίνσκ το 1992 ήταν ένα σημαντικό βήμα, αλλά το Αζερβαϊτζάν αρνήθηκε να εφαρμόσει ένα διεθνή μηχανισμό για την παρατήρηση των ε, παραβιάσεων της εκεχηρίας. Το Ναγκόφον Καραμπάχ έχει δημοκρατικούς θεσμούς, ένα υποδειγματικό δικαστικό σύστημα και χαμηλό επίπεδο διαφθοράς. Γι' αυτό το λόγο ε, ζητούμε τη συμπερίληψη εκπροσώπων του Ναγκόνο ε, Καραμπάχ στην ομάδα του Μίνσκ. Ε, αυτή τη στιγμή σε επιληθεί η στρατιωτική σύγκρουση θα μπορέσει να συμφωνηθεί μια διαδικασία ειρήνευσης ούτως ώστε να ενισχυθεί το νέο ανεξάρτητο κράτος. Επόμενος ομιλητής, ο κ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να σας πω ότι χάρη στους Ιταλούς δικαστές τώρα ε, έχει πέσει φως πάνω σε ένα καινούργιο σκάνδαλο όσον αφορά το ξέλιμα χρήματος σε σχέση με τα απορρίμματα και σε σχέση με τις, την ε, εξορρυκτική διαστηριότητα για εξέβρεση πετρελαίου στην Βασιλικάτα και αυτά τα έχουν και ε, πάρα πολύ αναμειχθεί αλλά και ο Πρωθυπουργός Ματιορέντζη 13 Νοεμβρίου ε, είπαμε, ε, είχαμε και συγκατάσταση εταιρεία ε, Τέμπα Ρώσα στις 7 Ιανουαρίου. Έχουμε διάφορες δραστηριότητε, κακές βιβλιοπτικέ για την υγεία και τότε έχουμε επίσης και καταστάσεις της ΕΝΗ που κάνουν εξόρυξη για πέμπτη φορά και επίσης έχουμε στη συνέχεια το ξέλμα χρήματο της Τεμπαρόσα και αυτά γίνανε με επίκεντρο το όλη τη Βιτζάνο και κατά αυτόν τον τρόπο εμείς ε, προσφύγαμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Το θέμα τι θα κάνουν οι ευρωπαϊκές αρχές γιατί όλα αυτά ε, γίνονται χωρίς να έχει υπάρξει κανένας είδους ε, ρύθμιση και κανόνας για να προστατεύσει την υγεία των πολιτών. Ο κύριος Μάριο Εγώ θέλω να καταγγείλω το ότι έχουμε μια πάρα πολύ σοβαρή παραβίαση των ε, προνομίων και αρμοδιοτήτων. Ε, κάτι το, στο οποίο έχουν προσφύγει επίσης και στο δικαστήριο του Μιλάνου. Ενώ από την νομική επιτροπή εξετάζεται το θέμα δεν θέλησε να αναστείλει την διαδικασία του το δικαστήριο του Μιλάνου. Επομένως τώρα παραβιάζεται πάρα πολύ η διαδικασία σχετική με το βουλευτικό προνόμιο αλλά έτσι παραβιάζεται και η πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και επίσης ε, απευθύνομαι και στον πρόεδρο Σούλς. Θα πρέπει ο πρόεδρος να προστατεύσει ε, τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητές μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν πρέπει να ανεχθούμε η αρχή της βουλευτικής ε, ελευθερίας γιατί περί αυτού πρόκειται ε, να καταπατάτε με τέτοιο κατάφορο τρόπο αλλά και να την πάγια νομολογία του ΔΕΚ. Ο επόμενος. Microphone, please doamnă președintă η κορίνα κρέτσου μέλος της επιτροπής juncker έχει κατηγορηθεί από συνεργάτες και δημοσιογράφους ότι δεν εκπληρώνει το έργο της, δεν πηγαίνει στο γραφείο της, μένει πολύ καιρό στη χώρα της ή με κάνει τις επίσημες επισκέψεις ιδιωτικές. Οι συνάδελφοι έχουν ζητήσει εξηγήσει φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να αποκρύψει αυτά ε, αυτά τα θέματα. Όλοι οι πολιτικοί συντάκτες έχουν γράψει για το, βιβλίο, για το φυλάδιο που δημοσίευσε σχετικά με, με, ευρωπαϊκά χρήματα. Ε, είναι ένα χαρακτηριστικό που ζήλευε και ο κύριος ε, Κατσαουσέσκο. Η κυρία Κρέτσου ε, έχουμε ζητήσει εξηγήσει για την κυρία Κρέτσο από την Επιτροπή και περιμένω να μάθω αν συμφωνεί ο κύριος Γιούρκερ ότι πρέπει ε, τα ευρωπαϊκά χρήματα να ε, δαπανώνται για ιδιωτικού λόγους τους Επιτρόπου. Ο κυριος Φερναντέ. Φερναντές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα, Α θυμηθούμε την λογιόλα τον, τον κύριο Παλάθιο, ο πυροσβέστης ο οποίος έδωσε τη ζωή του για να προστατεύσει ε, περιουσίες και ζωές στο Οβιέδο. Οπότε θα πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι με την οικογένεια αυτού του πυροσβέστη. Κοιτάξτε, θέλω να σας μιλήσω τώρα για τα γαλακτοκομικά στην Αστούρια. Πάνω από 2.000 οικογένειες τώρα έχουν ε, πρόβλημα, πρόβλημα επιβίωσης γιατί δεν υπάρχουν κάποια αποφασιστικά μέτρα από την Επιτροπή και το Συμβούλιο που θα εγγυώνται κάποιες εύλογες τιμές. Μέτρα παρέμβαση στην αγορά. Ο καταναλωτής να μπορεί να ξέρει πού προέρχεται το γαλακτοκομικό προϊόν. Να σταματήσει το dumping. Γιατί ο κλάδος τώρα βρίσκεται σε αδιέξοδο. Πρόκειται για αυτό το γάλα που είναι από την Αστούρια και αξίζει να το εξασφαλίσουμε το μέλλον λέει πίνοντας γάλα ο ομιλητής. Ευχαριστώ. Και τώρα κύριε Φωτού, Φωτούγκα. Φωτίγκα. Φωτίγκα, Φωτίγκα ονομάζομαι λέει. Στην ε, η περιοχή μου ήταν κατά της συμπεριαλιστικής πολιτικής της ε, Ρωσίας. Ε, η Γεωργία και η Ουκρανία θα πρέπει να προποθεθούν προειδοποιηθούν υπ' αυτή την έννοια. Αντιμετωπίζουμε μια αισχρή προπαγάνδα. Και διαρωτώ κατά πόσο αυτό δεν, έχει, δεν θα έχει κάποιο αντίκτυπο στο Ολλανδικό δημοψήφισμα. Οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υποστηρίζουν στο πλαίσιο της ε, κοινή ε, αμυντικής πολιτικής, πώς θα ε, αντιμετωπίσουν τις απειλές που προέρχονται από τη Ρωσία. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Σελίμοβιτς. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ράταν Κάρατζης ε, καταδικάστηκε για γενοκτονία και βεβαίως ε, δεν είπε την ε, αλήθεια. Και, μετά, και λίγες μέρες μετά από την απόφαση αυτή ο Σέσελη ε, αθώθηκε γιατί δεν μπόρεσε να διαπιστωθεί καμία σύνδεση μεταξύ της δικής του δραστηριότητας και των εγκλημάτων πολέμου. Βεβαίως ε, νομικά είναι δύσκολο ίσως να, αποδειχθούν αυτές οι, να αποδειχθεί αυτή η διασύνδεση. Δηλαδή ότι ε, για παράδειγμα έβγαλαν τα μάτια από τους ε, Κροάτες. Ωστόσο μια τέτοιου απόφαση είναι ανήθικη και θα πρέπει εμείς ως πολιτικοί να κάνουμε κάτι γιατί μια τέτοιου απόφαση έχει τεράστια επιπτώσει όσον αφορά την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να στυλιτεύσουμε ξεκάθαρα τέτοιου είδους εγκλήματα πολέμου και να πράξουμε σε ηθικό επίπεδο αυτό το οποίο παρέλειψε να κάνει το δικαστήριο της Χάη. Την προηγούμενη εβδομάδα λάβαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επίσκεψη ε, μαθητών που ζουν ε, κοντά σε δύο ε, εργοστάσια, σε δύο διελιστήρια πετρελαίου τα οποία έχουν, το ένα έχει κατασκευαστεί σε θαλάσσια περιοχή, το άλλο σε μια προστατευόμενη περιοχή φυσικού κάλους. Ε, οι περιοχές αυτές έχουν αυξημένα ποσοστά καρκίνων και πρόωρων θανάτου. Ε, θα πρέπει ε, οι κοινότητες ε, προτίμησαν να σπαταλήσουν τα κονδύλια για να υπερασπιστούν ε, αυτές τις βιομηχανίες αντί την υγεία των πολιτών. Ε, είναι απαράδεκτο να μην αντιμετωπίζετε τέτοιου είδου θέματα τα οποία επιβαρύνουν εξαιρετικά την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ, Λίκιο Σκρέτς. Τα νέα κράτη-μέλη, ιδίως στην Κροατία, από την οποία προέρχομαι, ε, ακόμα δεν ε, προβλέπουν κάποια μέτρα όσον αφορά την ανακαίνιση κτηρίων, Ιδίω όσον αφορά τι πιο δυνατέ κοινωνικέ ομάδε, δηλαδή διότι δεν προβλέπουμε τίποτα, δεν έχουμε νομοθεσία για την ενεργειακή παινία θα ε, πρέπει να δώσουμε κίνητρα για περισσότερη χρήση των ανανεώσιμων και έτσι να δημιουργήσουμε και θέσεις απασχόλησης. Η κυβέρνησή μας έδειξε ανευθυνότητα γιατί υποχρέωσε τους πολίτες να βάλουν κάποιους μετρητές όσον αφορά τα συστήματα θέρμανσης αλλά δεν τις και όταν καρφάκι όσον αφορά την ε, ανακαίνιση των ε, κτηρίων ούτε ενημερώθηκαν οι καταναλωτές για το τι τιμές θα έχει η θέρμανση που χρησιμοποιούν επομένως. Υπάρχει εδώ και νομοθεσία, αν όχι ε, παρανομία απλή, οπότε θα πρέπει κάτι να κάνει η Ευρωπαϊκή Ευρώπη για να προστατεύσει τους ε, συμπολίτε μου και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Microphone, please. Επιτρέψατε μου να σας ε, να αναφερθώ στα ε, σωστή θεωρεί η Τσεχία για την ε, συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Είναι κατά μια υποχρεωτικής ενός υποχρεωτικού συστήματος ανακατανομής. Είναι Δεύτερο, είναι κατά αυτού του συστήματος όσον αφορά τις ελαφρύνσεις για τους ε, πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο ενδιαφέρει καθόλου τις Βρυξέλλες αυτό το οποίο πιστεύει ένα δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιο. Όχι, θεωρώ ότι η Κομισιόν και το Συμβούλιο σκόπιμα προχώρησαν στη σύναψη μιας συμφωνίας με την ε, Τουρκία που δεν συνιστά επισήμω μια σύμβαση ακριβώς επειδή παρακάμπτει, επιθυμεί να παρακάμψει τα εθνικά κοινοβούλια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προέβησε μια τέτοιου είδους συμφωνία ε, επί της οποίας ε, δεν μπορούσε να αποφανθεί κανένα από τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν απολύτω καμία εμπιστοσύνη πλέον στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στις 6 Απριλίου οι Ολλανδοί αποφάσισαν με δημοψήφισμα να, να απορρίψουν τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Αυτό ήταν πρόσχημα. Αυτό το οποίο σκόπευαν οι πολίτες που ξεκίνησαν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διοικούντες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η αποτυχία της απέναντι στην μεταναστευτική κρίση. Έξι ηγέτες οι οποίοι συσσωρεύουν σκάνδαλα. Τα LuxLeaks, Panama Papers. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταλαβαίνει το μήνυμα που έχουν στείλει 64% των ψηφοφόρων. Αντί να διορθώσει την κατάσταση, ενισχύει ακόμα περισσότερο την τεχνοκρατικού δεσμού που πνίγουν τα κράτη-μέλη ας πούμε, τη δημιουργία ενός, μια Super Frontex για να σώσει το Schengen. Το Brexit 23 Ιουνίου περιμένουμε την, την, και την εμφάνιση της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία το 2017. Η κυρία Μαγκίνε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όχι για πρώτη φορά. Θέλω να μιλήσω εδώ στο χώρο αυτό για το εμπόριο και συγκεκριμένα το θέμα της ε, εμπορικής συμφωνίας με τις χώρες Μερκοσούρ. Ξέρω ότι στο Συμβούλιο Γεωργίας ε, στο Λουξεμβούργο σήμερα ακούστηκαν φωνές. 23 κράτη-μέλη ε, ανησυχούν για την τακτική σχετικά με το Μερκοσούρ για ευαίσθητα προϊόντα όπως το βόλιο κρέας αλλά και ε, το ε, και το κρέας πουλερικών. Ε, είναι σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει τις εισαγωγές βοήου κρέατος και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως τους αγρότες. Καθώς ακούστηκαν φωνές ε, στο Συμβούλιο Γεωργίας σήμερα το πρωί, ήθελα και εγώ να υψώσω τη φωνή μου και ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι συνέδελφοι της Επιτροπής Γεωργίας που ανησυχούν και θέλουμε να προειδοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην θυσιάσει τη Γεωργία προς χάρη άλλων τομέων της οικονομίας. Ευχαριστώ. Thanks. And next one... Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Τσάνι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχει διαμακρόν συζητηθεί αν, τα, κράτη, ε, αν θα πρέπει τα κράτη-μέλη ε, να έχουν δικά τους πρότυπα για την υπηκότητα ε, και την άδεια παραμονής. υπάρχει Ευρω οι πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα της ευρωπαϊκής υπηκότητας το έχουν θέσει υπό άλλη σκοπιά. Γιατί οι σοβαρές απειλές των τρομοκρατίας, το θέμα της ε, διαφυγής και η κρίση των προσφύγων έχει ε, δημιουργήσει πρόβλημα. Οι συνθήκες είναι δύσκολες, δεν υπάρχει διαφάνεια και άρα ε, εκεί αναπτύσσονται η απάτη, η διαφθορά και η τρομοκρατία. Κάποιες χώρες ανοίγουν σε ε, δίνουν τη δυνατότητα σε εύπορους πολίτες να, έχουν, να κινηθούν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά διευκολύνουν τόσο πολύ τους εύπορους να αποκτήσουν δικαιώματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άλλοι στην ουσία κινδυνεύουν την ίδια τους τη ζωή για να φτάσουν εδώ, στέλνουν και αυτό ε, το λανθασμένο μήνυμα. Το θέμα λοιπόν είναι θέλουμε να στηρίξουμε τη φοροδιαφυγή και να διατηρήσουμε την ε, άνηση, μεταχείριση των μεταναστών με βάση τα οικονομικά τους ή θα πρέπει να επιβάλλουμε αυστηρούς κανόνες και παρακολούθηση για να τα εμποδίσουμε αυτά. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κ. E, Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μιλάμε τώρα για ένα χωρίο του προημίου στην συνθήκη, οπότε θα πρέπει να αναζητήσουμε το αληθές νόημα και να μην θεωρήσουμε είναι απλώς διπλωματικό και διακοσμητικό, γιατί μιλάμε γιατί έχουμε τώρα την ε, χιλιοστή πεντηκοστή επέτειο της ε, ε, βαπτίσεως και αποφάνθηκε σε σχέση με αυτό και ο πρόεδρος του δικού μας κοινοβουλίου γιατί πριν 50 χρόνια είχαμε το ορόσημο, την χιλιαστή επέτειο. Η αυτή επέτειος σηματοδότησε την ελευθερία της Πολωνίας αλλά και άλλων εθνών στην Ευρώπη. Σήμαινε ότι θα υπάρχει ασφάλεια για όλους και επομένως βλέπουμε ότι η χριστιανική κληρονομία δεν είναι μόνο δική μας ε, κληρονομιά αλλά αποτελεί και μια ελπίδα για το μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το προσφυγικό βλέπουμε ότι κινδυνεύει να διαλύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορεί να εξασφαλίσει ασφάλεια ούτε μπορεί να καλύψει αυτές τις χιλιάδες των προσώπων που αξίζουν ε, προστασίας. Ε, έρχεται το ΝΑΤΟ και αναπτύσσει στρατιωτικές επιχειρήσεις, η Frontex, βλέπουμε την καταστολή και είδαμε τι έγινε εκεί μέσα στις λάσπες με τα αέρια που τους πετάξανε. Πάρα πολλά είναι τα λάθη και στην αντιτρομοκρατική πολιτική. Χρησιμοποίησαμε την, ε, τον βασανισμό και τώρα πετάμε στο καλάθι των αρχίστων τη σύμβαση της ε, Γενέβης. Μα ε, λέμε ότι είναι ασφαλής χώρα η Τουρκία, είναι εκεί ασφαλής η δημοσιογράφοι ή οι διανοούμενοι ή κανένας. Βλέπουμε πως χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες τους πρόσφυγες για να μας ε, εκβιάσουν και εμείς ε, τι κάνουμε, τους στέλνουμε σε ένα σφαγείο αυτούς τους ανθρώπους. Κυρία Σόντρου έχει το λόγο. Στις 17 Μαρτίου ε, συναντήθηκαν οι Υπουργοί Παιδείας στο Παρίσι και υπέγραψαν μια δήλωση για τις ε, κοινέ αξίες ε, της ε, ανεξιθρησκείας και των μη διακρίσεων στην εκπαίδευση ως αντίδραση στις επιθέσεις κατά του Σαλή Επτό. Ωστόσο θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί και βέβαια απειλούν και άλλα τρομοκρατικά χτυπήματα. Δεν ε, μπορούμε να αναμένουμε βεβαίως ε, θετικά αποτελέσματα, αλλά θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι οι προσπάθειες ένταξης ε, των ξένων στην γαλλική κοινωνία δεν τελεσφόρησαν. Γι' αυτό θα πρέπει να υποστηριχθούν τα εκπαιδευτικά συστήματα και να υπάρξει μια καλύτερη προετοιμασία των εκπαιδευτικών ούτως ώστε να διδάσκουν την ε, ανεξιθρησκεία και τις ε, σύγχρονες ευρωπαϊκές ε, δημοκρατικές αξίες. Ζίκα είναι μια παγκόσμια απειλή η πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι προκαλεί πολύ ευρύτερο φάσμα εγκεφαλικών παθήσεων από ό,τι αρχικά είχε θεωρηθεί. Ήδη έχουμε δει περιπτώσεις μικροκεφαλίας, γιγιομπαρές και άλλων προβλημάτων που ε, συνδέονται με αυτόν. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά εδώ και υπό την έννοια αυτή πρέπει να βελτιωθεί ο περιορισμός του ιού Ζήκα και να βελτιωθούν οι ερευνητικές μέθοδοι. Εδώ ο χρόνος πιέζει για τη διάγνωση αλλά και ε, για την εξέβρεση εμβολίου κυρίως για τις έγκες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που την προηγούμενη εβδομάδα είχε την επέτειό του έχει κάνει προσπάθειες να επιστηρίξει τις χώρες που πλήγονται από το Ζήκα. Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναφερθεί κρούσματα του ιού και αντιμετωπίζουμε το κίνδυνο μιας επιδημίας στην Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την περίπτωση αυτή. Πρέπει το ιατρικό προσωπικό να είναι σε επιφυλακή και ο, ο κόσμος να γνωρίζει τους κινδύνους. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής ο κύριος Τσαμπάσκι. Εγώ, συνάδελφε, θα ήθελα να σταθούμε στον εξισλαμισμό που αφορά τους Ρώμ της Βουλγαρίας. Πρόκειται για κίνδυνο κατά της κοινωνίας μας αλλά και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αποτέλεσμα όλες αυτής της διαδικασίας το νιώσατε και το νιώσαμε όλοι σε Βρυξέλλες και Παρίσι. Όλα αυτά παρά το ότι συνεχίζει η Τουρκία να κάνει αυτήν την σιωπηλή εισβολή στην Βουλγαρία. Πρόκειται για επιθετική πολιτική του Ερντογάν. Ήρθε η ώρα να καταλάβει η Ευρώπη τι απειλή αποτελεί η σημερινή τουρκική πολιτική. Πρόκειται για μια αυθεντική περίπτωση πολέμου. Αυτό κάνει η Τουρκία καθημών. Να σταματήσουμε να στρουθοκαμιλίζουμε. Ο επόμενος, Πολτσακ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η, τροπογρα... τρομοκρατία δεν γνωρίζει σύνορα, απειλεί την ελευθερία μας καθώς και την ε, ε, πίστη των σύνορα απλών ανθρώπων έναν των πολιτικών. Θα πρέπει να, έχουμε... να αποκτήσουμε νομικά εργαλεία στα χέρια μας ούτω ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους δράστες. Θα πρέπει να έχουμε το αίσθημα, να δείξουμε αίσθημα προσωπικής ευθύνης όσον αφορά τις τρομοκρατικές πράξεις. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μία νομική ρύθμιση ούτω ώστε τα δικαστήρια να μπορούν να τιμωρούν δράστες ε, τρομοκρατικών επιθέσεων με αφαίρεση της ηθαγένειας. Κατά την άποψή μου δεν είναι πλέον δυνατό οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, οι οποίοι ε, διαπράττουν ε, τρομοκρατικά δικήματα να διατηρούν την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Θα πρέπει να λήξει αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ Πρόεδρε Πίτροπε. Όλο και περισσότερες περιπτώσεις σεξουαλικής ε, ε, βίας από τα ε, άνδρες της ελληνικών δυνάμεων του ΟΗΕ συμπεριλαμβανομένων και στρατευμάτων που έχουν στείλει τα κράτη με της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται. Είναι φοβερό ότι οι πλέον ευάλωτοι του κόσμου αυτού, γυναίκες και παιδιά που έχουν χάσει τα πάντα, είναι άτομα που υποφέρουν από αυτούς οι οποίοι υποτίθεται ότι τους προστατεύουν. Έχω σοκαριστεί για αναφορές σε, σε περιπτώσεις κοριτσιών που αναγκάστηκαν ε, να κάνουν κτηνοδίες ε, από τους ε, τους στρατιώτες. Οι στρατιώτες οι οποίοι αναγκάζουν παιδιά να κάνουν σεξουαλικές πράξεις προκειμένου να τους δώσουν φαγητό. Αυτοί είναι άνθρωποι από όλες τις χώρες του κόσμου και η κατάσταση είναι αρρωστημένη. Ζητώ λοιπόν από την ύπατη εκπρόσωπο Μογκερίνη να θέσει το θέμα στην Ευρωπαϊκή, στο ε, ΟΗΕ έτσι ώστε όλοι αυτοί να, να... να διωχθούν ποινικά και να εξασφαλιστεί ότι τέτοιου τέτοιου είδου ε, καταχρήσει δεν γίνονται ανεκτέ. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ο κύριο uh, Κυρία Πρόεδρε, οι ε, εργαζόμενοι στον τομέα της χαλιβουργίας ε, και οι οικογένειές τους ανησυχούν για την παρούσα κατάσταση του, της χαλιβουργίας του Ηνωμένου Βασίλου. Βεβαίως βρέθηκε αγοραστής, αλλά χιλιάδες θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό που είναι σημαντικός για την ασφάλεια και την άμυνα του Ηνωμένου Βασιλείου τίθενται σε κίνδυνο. Η πρέπει να ξεκαθαριστεί ένα σχέδιο για τεσσάρων σημείων για την Χαλιβουργία και να ε, ε, γίνει ε, έρευνα σε διάφορο, στα διάφορες φάσεις. Επίσης έργα υποδομής, να ξεκινήσουν έργα υποδομής που χρειάζονται μεγάλες ποσότητες χάλιβα. Πρέπει να υπάρξει ενδιαφέρον για το μέλλον της Βρετανικής χαλιβουργίας. Τώρα πρέπει να υπάρξει ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα και να υπάρξει απαγόρευση της εισαγωγής φθηνού κινέζικου χάλιβα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάρα πολύ θετικά είναι τα ε, σημερινά νέα ότι αυτή η βιομηχανία ε, βοήθησε το Σκάνθρωπ διασώθηκε η τοπική εταιρεία, η τοπική χαλιβουργία. Τελικά είναι ε, θέμα ύπαρξης της βιομηχανίας μας με όλο αυτό το dumping γιατί βλέπουμε ότι αντίθετα με αυτό που λένε οι ευρωσκεπτικιστές η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει με τέτοια ε, εμπορικά μέτρα αμυντικά. Μιλάμε για 72% του πληθυσμού της Ευρώπης που είναι υπέρ ανάληψης δράσης ε, από την Ευρώπη αλλά τελικά η δική μας κυβέρνηση εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει οπότε είναι εδώ σε κάποιες εβδομάδες να ξεμπλέξουμε όλα αυτά. Ε, το Μάιο έχουμε το σχετικό συμβούλιο και εάν θέλει ο Κάμερο να σώσει τη χαλιβουργία μας, ξέρετε να κάνει. Και τώρα ο κύριος Μανίκινς. Πρόεδρε, κάθε κράτος δικαιούται να προστατεύει τους κατοίκους την ιδεφική ακυρότητα, τα συμφέροντά του με όποια μέσα είναι πιο πρόσφορα για το επιθυμητό αποτέλεσμα και μεταξύ αυτών των σημαντικών στοιχείων είναι η ελευθερία της γλώσσας, βασικές ελευθερίες και αυτός ο συμπατριώτης μας κατά σε φυλάκιση έξι μηνών κατά της του λόγου. Και ακόμα χειρότερα το Κοινοβούλιο τροποποίησε το ποινικό δίκαιο. Οπότε απαγορεύονται ακόμα και κάποια αστεία. Και τώρα ακόμα και κάποιες εκφράσεις, κάποια αστεία επιδέχονται φυλάκιση. Ε, ντρεπόμαστε για αυτά τα οποία έκανε η κυβέρνησή μας. Σας ευχαριστώ. Πρόκειται για τον τελευταίο ομιλητή. Συνεχίζεται η Ολομέλεια αύριο στις 12 Απριλίου του 2016. Είναι με 2.30 και 3 η ώρα με 11. Μπορείτε να βρείτε στο website του Ευρωκοινοβουλίου την ημερησία διάταξη. Πέρα στη συνεδρία σας. Τουλκέιλε. Ja,